λάβαμε 7 σχέδια ψηφίσματος. Η ψηφοφορία θα γίνει αμέσως μετά τις συζητήσεις. Τελειώνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Σαουδική Αραβία και η περίπτωση του Ραϊφ Μπαντάουι. Λοχ Μπίλερ για ένα λεπτό. το γεγονός πως αναβλήθηκε πολλές ε, φορές ε, ο δημόσιος βασανισμός του Ραΐφ ε, Μπαντάου για λόγους υγείας δείχνει τι τραγικά αποτελέσματα έχει η δημόσια μαστίγωση. Ποιος ξέρει τι θα γίνει με τους επόμενους 950 αραβδισμούς. Ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή του. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Πάρα πολλοί άνθρωποι συλλαμβάνονται, δεν υπάρχει δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης. Πέρσι εγώ συνάντησα τον δικηγόρο του κυρίου Μπαντάου, τον κύριο Αλκαΐρο, ο οποίος επίσης καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση. Εγώ προτείνω η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει έναν κατάλογο όλων των μη βίαιων πολιτικών κρατουμένων και να εγείρει αυτό το ζήτημα συνεχώς. Σας ευχαριστώ. Ντέμες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αποκτήσει ένα διπλωματικό βάρος. Το 2016 θα αποκτήσει έδρα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και μας λέει πως καταπολεμά την τρομοκρατία. Μπορεί λοιπόν η Σαουδική Αραβία να κερδίσει με το να καταδικάσει ρητός το Ισλαμικό κράτος. Βλέπουμε πως υπάρχει όλο και περισσότερη αναφορά στα μίμιε για το θέμα αυτό και ένα βήμα ανανέωσης νομίζω μπορεί να ωφελήσει τη χώρα των δύο Αγίων Τόπων του Ισλάμ αλλά βεβαίως κάτω από την επιφάνεια έχουμε ένα βάναυσο σύστημα το οποίο τιμωρεί τους ανθρώπους για επαφή με άλλες θρησκείες ε, και αποκεφαλίζει δημοσίως ε, λαθρεμπόρους, ε, μιχούς και λοιπούς. Παρουσιάζεται η χώρα ως σύγχρονη, αλλά στο εσωτερικό βρίσκεται στον Μεσαίωνα. Ελπίζω η Ευρώπη να είναι ενωμένη και να ξεκαθαρίσει η Σαουδική Αραβία πως δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ χωρίς να κάνει τίποτα στο εσωτερικό της. Ο Ραΐφ Μπανταούι δεν πρέπει να είναι φυλακή, αλλά σε ένα πάνελ τηλεοπτικό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σχάκε, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ο blogger Σαουδική Αραβία Μπαντάουι δεν ε, είναι σε θέση, σε φυσική κατάσταση για άλλους ραβδισμούς μετά τους πρώτους 50 που έλαβε. Οι ίδιοι γιατροί δηλαδή επιβεβαιώνουν πόσο βάρβαρη ήταν η μεταχείριση αυτή που βέβαια αντιτίθεται σε όλες τις συμβάσεις που η ίδια η Σουδική Αραβία έχει συνυπογράψει. Υπό το φως λοιπόν των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σουδική Αραβία εναντίον όλων των πολιτών αλλά κυρίως των γυναικών και όσων επικρίνουν το σύστημα το να είναι μέλος στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ΙΕ ειλικρινά είναι κοροϊδιά. Δυστυχώς όμως και στο σώμα αυτό είναι δύσκολο να μιλήσουμε με μία φωνή όσον αφορά την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Δική Αραβία. Και ζητάω από όλα τα πολιτικά κόμματα να υποστηρίξουν το κοινό ψήφισμα αυτό οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος του Μπανταούι πρέπει να καταδικαστούν με μία φωνή από όλου μας. Και ήρθε η στιγμή πια να σκεφτούμε ποιες είναι οι σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι μια αξιόπιστη, ένας αξιόπιστος σύμμαχος τη στιγμή που εξάγει φονταμεταλισμό, ακραίες θέσεις εδώ και όνες και χρησιμοποιεί την ίδια σκληρή βία όπως αυτή της τιμωρίας που εμείς τόσο πολύ καταδικάζουμε και που εφαρμόζει και το Ισλαμικό κράτος που εμείς καταδικάζουμε. Ευχαριστώ. Κοράω τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Ράφι Μπεντάβη, ε, μπλόκερ, και ήταν ο ιδρυτής των φιλελευθέρων σε όλοι συμφωνούμε τι γίνεται και γι' αυτό και θέλουμε αυτό το ψήφισμα για να απαιτήσουμε από τις αρχές Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσουν την ε, ποινή του και να τον απελευθερώσουν. Όμως θα πρέπει να μας προκληθεί ένας άλλος προβληματισμός ευρύτερος. Τι γίνεται με τα πετροδολάρια, τι σχέσεις έχουμε εμείς με τη Σαουδική Αραβία. Γιατί τώρα μιλούμε για συνεχείς καταπατήσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με μια χώρα που είναι σύμμαχος της Δύσης. Οπότε και δημιουργείται μια υποκρισία όταν μιλάμε για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μιλάμε για το Ισλαμικό κράτος από την άλλη μεριά. Έχουμε τέτοιες ίδιες πρακτικές σε μια χώρα φίλη. Έχουμε τέτοιες ποινές ε, ε, σωματικές σε όποιον επικρίνει το καθεστώς. Αυτή είναι η σκέψη μου. Ευχαριστώ κύριο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για απερίφραστη καταδίκη που πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την μεταχείριση του κυρίου Μπαντάουι. Χίλιες, ε, χίλιες φορές μας και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια, οπότε θα πρέπει να δούμε ότι εκεί υπάρχει θανατική ποινή στη χώρα αυτή, ποια είναι η θέση της γυναίκας, ποια είναι η θέση των ε, δυτικών ηγετών όσον αφορά την καταδίκη του Σάντραβ. Η κυρία Μέρκελ λέει για το ελληνικό χρέος και όμως ο Ντέβιτ Κάμερον είπε ότι θλίβει πάρα πολύ για το θάνατο του φύλακα των ε, τζαμιών. Επίσης ε, εξέφασε ελληνική και ο Μπαμ. Άρα εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άλλη στάση έχουμε με τους ισχυρούς και άλλη με τους αδύνατους. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, ότι, έτσι στηρίζονται οι, οι εξτρεμιστές Ένα μισό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι δικαστές οι οποίοι καταδίκασαν τον Ραϊφ Μπαντάουι σε δεκαετή φυλάκιση και εραυσμούς δεν είχαν ιδέα το τι προκάλεσαν. Ήταν μία από τις πολλές καταδίκες ε, πολιτών της Σαουδικής Αραβίας που απλά εξέφρασαν τη γνώμη τους. Όμως αυτή η περίπτωση έγινε γνωστή παγκοσμίω. Και πραγματικά μετέδωσε σε όλο τον κόσμο τις φρικτές σωματικές ποινές που επιβάλλονται στην Σαουδική Αραβία με μαστιγώσεις ε, καθεκάστην. Όταν το κάνει αυτό μια τρομοκρατική οργάνωση, δικαίω λέμε πω είναι κάτι το απεχθέ. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια, με μια χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε έντονα στον οικονομικό τομέα και μα συνδέουν συμφέροντα στον τομέα τη ασφάλεια. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να δεχόμαστε τέτοιε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σταθερότητα στην περιοχή δεν θα εξασφαλιστεί άμα κάνουμε τα στραβά μάτια μόνο μέσω της δημοκρατίας και ενός συστήματος δικαιοσύνης σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει μία μπλε κάρτα. Την δέχεστε από τον κύριο Βάγγελ. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, στην ομιλία σας αναφέρατε και την δυσκολία που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην όλη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε πολλές χώρες όπου παραβιάζονται τέτοια δικαιώματα. Το Ισραήλ, το Μαρόκο και άλλες και όλες ε, φιλικές τις θεωρούμε, εταίρους ε, και τα λοιπά. Έχουμε συμφωνίες. Ε, δεν νομίζετε πως έχει φτάσει η ώρα στο κοινοβούλιο αυτό να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το τι κάνουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια πολιτική στο μέλλον. Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματικά είναι αυτοτελή και δεν μπορεί να συνδέονται με άλλα ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες οι οποίες ε, αλλού μας κάνουν να ε, μιλούμε και αλλού να σιωπούμε. πρέπει πράγματι να είναι πέρα από τα πολιτικά συμφέροντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριος Πρέντα για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, οι αρχές της οδικής αραβίας ε, προχώρησαν σε ραβδισμούς σε βάρος του κύριου Μπανταουιέ. Η ελευθερία εκφρασής δεν μπορεί να τιμωρείται. Δεν συμφωνήσαμε με το ψήφισμα των άλλων ομάδων γιατί το κοινό ψήφισμα δείχνει ότι βάζει επί ίσες ώρες το Ισλαμικό κράτος και τη Σαουδική Αραβία μέσα σε μία και την ίδια παράγραφο. Είναι σφάλμα αυτό. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πάει αύριο στο ΡΙΑΤ. Οι συνάδελφοι δηλαδή, τι είναι σαν να πηγαίνουν στο Ισλαμικό κράτος, ονειρεύομαι. Και συγγνώμη δηλαδή που βλέπω ότι οι δύο προτάσεις έρχονται από το ΕΛΚΑ που είναι την Νάντια Σαφτσένκο και για τους Τατάρους στην Κρυμαία που διώκονται από τη Μόσχα αυτή την εποχή είναι δύο υποθέσεις που κρίθηκαν ότι δεν έχουν καμιά σχέση με το θέμα. Ευχαριστούμε Κέλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η περίπτωση του Ρεϊφ Μπανταουή πρέπει να προσεχθεί όλος ιδιαίτερος γιατί κανείς δεν μπορεί να φυλακίζεται και να τιμωρείται τόσο αυστηρά επειδή εκφράζει απόψεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. είναι μια απόφαση απαράδεκτη για μας. Η Σεουδική Αραβία εξάλλου έχει υπογράψει τις συμβάσεις κατά των βασανισμών. Συνεπώς απαγορεύονται οι βασανισμοί εκεί. Ελπίζω η συζήτηση αυτή να πείσει τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσουν την καταδίκη αυτή για ραβδισμούς και γενικά τις κατηγορίες σε βάρος του κύριου Μπανταουή και να του προσφέρουν ανθρώπινη μεταχείριση. Συγχρόνως, χαιρόμαστε για τις κάποιες μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη αρχίσει στην Σαουδική Αραβία και ενθαρρύνω τον νέο βασιλιά να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους πολίτες. Ευχαριστούμε, Ρίτσαρτ Χάουιτ. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, ραπτισμοί είναι βασανισμός και ο βασανισμός είναι κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία, ελεύθερη έκφραση και όχι παραβίαση τέτοιων δικαιωμάτων. Χίλιοι ραβδισμοί σε βάρος του Ραΐθ Μπανταουί... είναι κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλοι νιώθουμε τον πόνο από τους ραβδισμούς αυτούς και όλοι πρέπει να αντιδράσουμε. Η σύζυγος Σαφάρη λέει ότι υποφέρει τόσο πολύ που δεν μπορεί να μιλήσει για αυτό το θέμα και το μόνο που μπορεί να πει είναι πόσο βασανίζονται και τα παιδιά τους από αυτήν την απόφαση. Πρέπει να μπορέσει να βρεθεί με την οικογένειά του. Εμείς αυτό ζητάμε. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα είπε συνεργασία με τη Σεουδική Αραβία όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, μην ξεχνάμε ότι από εκεί έχουν βγει διάφοροι τρομοκράτες η για τη Σαουδική Αραβία αν πρέπει να σημαίνει κάτι αυτό, πρέπει να υπάρχει και ελευθερία, ελεύθερη ζωή στη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε. Χένκελ. Ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται πως η περίπτωση Μπαντάου είναι χαρακτηριστική περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας. Ήμουν μέλος ε, επί σειρά ετών ε, της ε, Διεθνούς Αμνηστίας ε, και μας λένε εδώ πέρα πως δεν έχει σχέση με το Ισλάμ. Διαχωρίζουμε το Ισλάμ από τον Ισλαμισμό σαν να διαχωρίζαμε τους σοσιαλιστές από τον σοσιαλισμό ή το κεφάλαιο από τον καπιταλισμό. Κι όμως σε 55 χώρες αυτή τη στιγμή παραβιάζονται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη να αντιμετωπίζονται οι γυναίκες διαφορετικά από τους άντρες. Τα περισσότερα θύματα είναι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό θεωρώ πως θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ε, όλες τις μουσουλμανικές χώρες. Ο κ. Χόλτερ έχει δίκιο. Δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σας ευχαριστώ, Ντεπρέ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αφόρητο, είναι τραγικό ε, αυτό το που έγινε με τον κύριο αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτό δεν είναι μία απομονή περίπτωση. Πρόκειται για ε, συνεχή καταστολή. Είναι αφόρητο γιατί πρόκειται για ένα ολόκληρο σύστημα. Και το χειρότερο είναι ότι πρόκειται για ένα σύστημα δικαϊκό, το οποίο το φτιάξανε και το ενεργοποίησαν οι, τα θεσμική φορή μια χώρας που τη θεωρούμε σύμμαχο. Και το ακόμα πιο τραγικό και αφόρητο ε, αυτής της ποινής που στον κύριο Μπαντάβη δεν είναι μόνο τη βαραυσότητα των ραβδισμών, είναι το ότι κατηγορείται για προσβολή του Ισλάμ ενώ αυτός απλώς χρησιμοποιεί το ε, ίντερνετ ούτως ώστε να κινητοποιεί έναν δημοκρατικό διάλογο. Επίσης είναι τραγικό το ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του τι κάνει το Ισλαμικό κράτος που βομβαρδίζουμε και από την άλλη μεριά τη πολιτική αυτή θεμητή και νόμιμη της Σαουδικής Αραβίας στην οποία και υποστηρίζουμε. Παρακαλώ όλοι οι συνάδελφοι να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία. Ε, Άλιν Σμιθ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουμε υποχρέωση προς τους λαούς όλες αυτές τις περιοχές ε, και δεν έχουμε αναγκαστικά ε, κάποια δέσμευση προς το καθεστώς το οποίο θα αλλάξει. Εγώ έχω έναν φίλο που μεγάλωσε στο Ριάντ και πέρασε για χρόνο μαζί του και έχω πολλές καλές αναμνήσεις και επομένως θα πρέπει να είμαστε πιστοί στις αρχές μας και άρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτή τη συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία από πλευράς της Σκοτίας έχει κάνει πολλά και ήταν πάρα πολύ σημαντικός και αποφάσισαν γι' αυτό να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή οι αρχές της χώρας. Αλλά έχουμε και άλλες περιπτώσεις ε, τέτοιες και άρα θα πρέπει το ψήφι να αφορά όλους αυτούς όπως και ο κύριος Χάουιτ. Εάν η συνεργασία με μια χώρα σημαίνει κάτι θα πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει να συμμορφωθούν με αυτές τις αρχές, αυτές οι χώρες. Να σκεφτόμαστε λιγότερο το εμπόριο των όπλων και να σκεφτόμαστε περισσότερο στο Βασίλειο για τι. Ε, ε, αρχές μας. Κασφάλτο ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χίλιοι ραβδισμοί για κάποιο είδους ε, blog που είχε θέματα θρησκευτικά και δημοκρατικά και πρόκειται για κάποιον ο οποίος ήθελε να παρασυρθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ε, πρόκειται για μια αργή καταδίκη σε αργό θάνατο. Επομένως, ε, τι να πει κανείς ο πολιτικής για τέτοιο βαρβαρισμό. Πρόκειται για μια χώρα που είναι εταίρος μας, η οποία θα όφιλε να ακούσει αυτό το οποίο λέμε και θα έπρεπε να ε, απελευθερώσει αυτούς που υποφέρουν έτσι. Θα πρέπει να αναθεωρήσει το ποινικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να φερόμαστε σαν τον χαμελέοντα και, και να φερόμαστε τέτοιο διαφορετικό τρόπο προς κάθε χώρα. Δεν είναι δυνατόν να ξεπουλάμε τις ε, αρχές μας εις όφελος του εμπορίου του πετρελαίου. Ο ραβδισμός του Μπαντάουι είναι μαστίγωση προς εμάς, προς όλη την Ευρώπη, προς τις αρχές μας. Και άρα οφείλουμε να κάνουμε κάτι προς τον ΡΑΙΦ και όλους τους άλλους ΡΑΙΦ που κρατούνται εκεί. Να χρησιμοποιήσουμε παν μέσων που διαθέτουμε και θα πρέπει να ενωθούν για αυτό όλες οι πολιτικές ομάδες. Δέχεστε. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Ωραία. Κύριε Καστάλτο. Μετά από αυτά που έγιναν στο Παρίσι μετά από τρομοκρατική τι επιθέσεις κατά του Σαρλί Εμπτό ο πρέσβης της Σαουδική Αραβίας στην Γαλλία παρέστη, συμμετέσχε εις την διαδήλωση όλων αυτών των προσωπικότητων που ήταν αλληλέγγυοι προς το Σαρλί Εμπτό και έστειλε αυτό το αντιτρομοκρατικό μήνυμα ταυτόχρονα έγιναν όλα αυτά στη Σαουδική Αραβία και εάν ε, είχαν γίνει όλα αυτά, αν υπήρχε σάλιμπτο δηλαδή στην Σαουδική Αραβία, ε, τότε οπωσδήποτε θα είχαν επιβληθεί τιμωρίε, ε, θανατικέ ποινέ, ε, χίλιοι ραβδισμοί κλπ. κλπ. Οπότε και ξεκίνησε ένα καινούριο κίνημα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διακόπτει ο πρόεδρο. νομίζω υπάρχει ένα τέτοιο κίνημα ε, όπω με το σύνθημα ή Σαρλί. Είμαι Σαρλί, εμπλό. Ναι, ναι, συνάδελφε, 100% σύμφωνα μαζί σα. Όχι, δεν πρέπει να αποδεχθούμε τέτοιου είδου ε, υποκριτική συμπεριφορά. Εάν θέλουμε να καταπολέσουμε την ε, τρομοκρατία, τότε θα πρέπει αυτό να το αποδείξουμε και θα πρέπει να ισχύσουν οι αρχέ μα, να, να, αποστασιοποιηθούμε από τέτοιε βαρβαρική συμπεριφορά. Θα πρέπει και εμεί κάτι να, κάνουμε. Οπότε συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε. Ε, ε είμαι ε, ραΐφ. Είμαι ραΐφ κάθε μέρα. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Πρόκειται οπωσδήποτε ο κύριος Κέλλη για μια πολύ θλιβερή περίπτωση. Γιατί από τη μια μεριά έχουμε αγαστές σχέσεις με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και έχουμε ολόκληρη συμφωνία εταιρικής σχέσης αλλά από την άλλη μεριά έχουμε μια χώρα, ένα βασίλειο, το οποίο φημώνει τις φώνες που στο καθεστώς, αλλά αυτό είναι αφόρητο, δεν είναι δυνατόν αυτό να το ανεχθούν. Επομένως, θα πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε τέτοιου παιχνίδια και θα πρέπει να καταβάλουμε πάσα δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να ασκήσουμε πίεση προς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για να μπει ένα τέλος σε αυτού του είδους τις ε, βαρβαρικές ενέργειες. Και θα πρέπει να πιέσουμε για να απελευθερωθεί ο Ράιφ. Η κυρία Βαλεντιάνο. Ευχαριστώ. Σαουδική Αραβία. Χώρα εταίρος. Μπανταουί. Μπλόγκερ. Δέκα χρόνια φυλάκιση, χίλιοι ραβδισμοί, βασανιστήρια και θάνατος. Οι διεθνείς οργανώσεις απαιτούν την απελευθέρωσή του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να περάσει ένα κοινό μήνυμα. Γιατί το ΕΛΚ δεν θέλησε να συμφωνήσει και να συνυπογράψει μαζί μας το κοινό ψήφισμα. Αυτό είναι ένα παραπάνω βασανιστήριο για τον Πανταουή. Οι ηγέτες των ε, κυβερνήσεων, οι πρέσβεις, οι διπλωμάτες, οι επιχειρηματίες που πηγαίνουν σε Οδική Αραβία δεν θα πρέπει να μπορούν να μιλήσουν για τα Πανταουή. Ελπίζουμε ότι όλοι αυτοί οι φάκελοι που θα φτάσουν σε οδική Αραβία, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίε, οι πολιτικοί κτλ. που θα πάνε εκεί, να βρουν λίγο χώρο στι τσάντε του να βάλουν και κάτι για τον Μπανταουί. Αλλιώ θα έχει μείνει με το στόμα κλειστό Ευρωπαϊκή Ένωση. Catch the eye. Τώρα. Παρακαλώ, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δύο μόνο θα μιλήσουν στη διαδικασία αυτή. Catch για να κερδίσουμε κάπως χρόνο. Αυτό σημαίνει ο κύριος Μοτεμπέλη έχει το λόγο πρώτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή για τη Σαουδική Αραβία είναι μια καλή ευκαιρία για να θέσουμε τα πραγματικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, βρίσκουμε φυσιολογικό η χώρα αυτή να μην αναφέρεται ποτέ στα κατεπήγοντά μα, ενώ πολλέ φορέ θα έπρεπε να αναφέρεται. Έπειτα υπάρχει ο δημοσιογράφο, ο blogger, ο Μπανταουή, για τον οποίο μιλάμε σήμερα, που έχει καταδικαστεί 10 χρόνια φυλάκιση, χιλιραυδισμοί. Γιατί, γιατί απλώ έκανε τη δουλειά του ω δημοσιογράφο. Και εδώ θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Λαγκάρτη, πρόεδρο ε, του Δούνου του, που εξέφρασε την θλίψη του για το θάνατο του βασιλιά, ο οποίο είχε κάνει πολλά για τι γυναίκε. Ναι, ναι, δεν είναι αστείο. Από εκείνη η Βυρμανή, άλλοι δύο γυναίκε στη φυλακή εδώ και χρόνια, γιατί τόλμησαν να οδηγήσουν αυτοκίνητο στη χώρα. Ο Ραϊφ Μπανταουή λοιπόν τιμωρείται για όλους αυτούς άντρες και τις γυναίκες που το μόνο που κάνανε ήταν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν μπορεί λοιπόν να διαδηλώνουμε για να κάνουμε κάνουμε για το Σαρλίκα από την άλλη μεριά με τα πετροδολάρια να σιωπούμε. Η κυρία Νότσεκα ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι υπάρχει πλειοψηφία έξι κοινοβουλευτικών ομάδων που ζητάνε την άμεση και να απελευθέρωση του κυρίου Μπαντάουι. Γιατί ο ραβδισμός είναι βασανιστήριο και τα δέκα χρόνια φυλάκιση για την έκφραση γνώμης είναι βάρβαρη ποινή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε. Και αναρωτιέμαι πραγματικά γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με όλη, δεν συμμετέχει σε αυτή την αλληλεγγύη. Μα γιατί πραγματικά δηλαδή το πετρέλαιο είναι σημαντικότερο από τον αγώνα κατά της βάρβαρης παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλλον αυτό θα είναι. Αυτή η έλλειψη αλληλεγγύης πραγματικά είναι κάτι το οποίο καταδικάζω και χαίρομαι για αυτό το οποίο καταφέραμε χωρίς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καταδικάσουμε δηλαδή αυτούς τους ραβδισμούς. Να πω κάτι για την Αυστρία περιμένουμε ακόμα επιτέλους να ζητήσει το κέντρο Αμπτουλάχ στη Βιέννη την άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση του Ραΐφ Μπαντάουι. Λευτεριά στο Ραΐφ Μπαντάουι. Τον λόγο έχει ο Επίτροπος ο κύριος Στυλιανίδης. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Στυλιανίδης, αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα για την υποστήριξή σας, γιατί θα ε, επιψηφίσετε την προσπάθειά μας ούτω ώστε να εφαρμοστούν παντού σε όλο τον κόσμο τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί η Σαουδική Αραβία είναι ένα σημαντικό εταίρος για την Ένωση. Είναι μια χώρα που επηρεάζει σημαντικά πολιτιστικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, ε, το γίγνεσθε στην Μέση Ανατολή και στον Ισλαμικό κόσμο γενικότερα. Και πάρα πολύ προβληματιστήκαμε εδώ στην Ευρώπη από την ποινή που επευλήθη στον κύριο Μπανταουή. Έγινε αυτό από το Σαουδικό ε, εφετείο τον Σεπτέμβριο πέρσι και έγινε επίσης δημόσιος ε, ραβδισμός του ε, που ξεκίνησε στις 9 Ιανουαρίου φέτος και με προσοχή παρακολουθούμε τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με αυτή την υπόθεση αλλά και παρακολουθούμε το τι γίνεται με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Αναμφίβολα. η ποινή του, το είδος της ποινής που επιβλήθηκε, μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Επίσης, αυτή η ποινή είναι κατάφορα δυσανάλογη. Επίσης, είχαμε την ε, ανακοίνωση της Φεντέργα Μογκυρίνη, της υπάτης εκπροσώπου, τον Ιανουάριο και υπενθύμησε ποια είναι η ακλόνητη θέση μας για το γεγονός αυτό. Πρόκειται μόνο για μία από τις περισσότερες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεχώς παρακολουθεί τις εξελίξεις της υπόθεσης και μέσω της αντιπροσωπείας μας στο Ριάντ. Συντονιζόμαστε με πολλά κράτη-μέλη για διάφορες ε, επίσημες και ανεπίσημες ενέργειες και επαφές που γίνονται με τη Σαουδική Αραβία και στις ε, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στην χώρα την ίδια. Είχαμε πρώτα-πρώτα στις 9 Ιανουαρίου 50 ραβδισμούς και ε, στη συνέχεια όμως ανεστάλλει εκτέλεση της ποινής για λόγους υγείας. Αυτό ήταν μια θετική εξέλιξη. Οπότε και ελπίζουμε ότι η εκτέλεση της ποινής δεν θα γίνει. Και εμείς θα συνεχίσουμε τις εκκλήσεις προς τους ε, Σαουδάραβες εταίρους, τόσο ώστε να ε, αναθεωρήσουν την απόφαση αυτή του δικαστηρίου και να αναπαινθεί και πάλι η απόφαση στο εφετείο γενικότερα αυτό το οποίο θέλουμε να ξεκινήσει ένας ειλικρινής διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους ε, φίλους Σαδάραβε. και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μια ευκαιρία ούτως ώστε και εκείνοι να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό του σύστημα και να καταργήσουν τις ε, σωματικές και ταπεινωτικές ποινές να εξεταστεί ευρύτερα το θέμα της ελευθερίας, της έκφρασης κάτι το οποίο είναι πάλι βασικό στοιχείο για τον διάλογο ημών και εκείνων. Οπότε και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με προσοχή την υπόθεση Μπανταουή. Θα συνεχίσουμε να στέλνουμε αυτό μας το μήνυμα από τους κατάλληλους διάβλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Πίτρο Πρόεδρος. Τώρα, έχουμε 7